Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι έκθεση του κύριου Μπουτικόφερ, αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη. Είναι το θέμα της έκθεσης. Δίνω ευθύς αμέσως τον λόγο στον κύριο Μπουτικόφερ. Πείτε. Κύριε Αντιπρόεδρε, εξάρτημε συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις στην Επιτροπή Βιομηχανίας και τους συναδέλφους από πολλές άλλες επιτροπές που συνεργάστηκαν μαζί μας, ιδιαίτερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, την Επιτροπή, αλλά και πάρα πολλούς φορείς από την κοινωνία των πολιτών. Πράγματι, η πολιτική για τις πρώτες ύλε είναι μία από τις μέζονες προκλήσεις για τη βιομηχανία, αλλά ταυτόχρονα είναι μια, μια τεράστια ευκαιρία. Εγώ τον τελευταίο 1,5 χρόνο ασχολήθηκα ιδιαίτερα με αυτό το θέμα. Με αφορά ιδιαίτερα και είμαι πεπισμένος πως ε, με μία προσεκτική μεν αλλά φιλόδοξη στρατηγική καινοτομία. Ε, ε αντιθέσιμο στο επίκεντρο των προσπαθειών μα θα έχουμε μεγάλη επιτυχία. Αποδοτικότητα των πόρων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση αλλά και υποκατάσταση. Αυτέ είναι σημαντικέ στρατηγικέ περί των οποίων πρόκειται εδώ ε, και ε, θα πρέπει τη μελλοντική μας ανταγωνιστικότητα να στηρίξουμε ακριβώς αυτή τη ε, στρατηγική καινοτομία. Ε, δεύτερον, εάν θέτει κανείς κάποιους στόχους αλλά δεν σκέφτεται τα εργαλεία για να τις επιτύχει, σπάνια μπορεί κανείς να πετύχει κάποιον από αυτούς τους στόχους. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε το ζήτημα αυτό και να ε, ε, δούμε ξεκάθαρα το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ των χωρών μελών ή μεταξύ χωρών μελών και επιτροπής να οργανώσουμε πολύ καλά αυτή τη συνεργασία. Μία αποτελεσματική διακυβέρνηση είναι, ε, έχει το ρόλο κλειδί για την επίτευξη αυτού του θέματος, του στόχου. οι, πρώτε, οι ορυκτές πρώτες ύλες είναι ιδιαίτερα σημαντικές όπως το πετρέλαιο, το αέριο, ή άλλοι ενεργειακοί πόροι. Αλλά μέχρι στιγμής δεν διαδραματίζουν ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο και εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Και σε αυτή την έκθεση αναφέρουμε μια σειρά από εργαλεία μέσω των οποίων μπορούμε να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση, την governance. Ένα σύστημα ραντάρ κινδύνου, ένα κατάλογο για τις κρίσιμες σημασίες πρώτες ύλες ε, ε, όπως το λίθιο για παράδειγμα ε, που ακόμα δεν έχει συμπεριληφθεί στο κατάλογο είναι στρατηγικής σημασίας. Προτείνουμε επίσης ένα δίκτυο αρμοδιοτήτων για τις σπάνιες γέες. θα υπέρ ε, η πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια σύναψη εταιρικές σχέσεις με στόχο την αποδοτικότητα των πόρων να προωθηθεί. Ε, θέλουμε οι διάφοροι δρόντες, οι γενικές διευθύνσεις, τα κοινά ερευνητικά κέντρα, ε, οι ξένες διπλωματικές, η ε, εξωτερική υπηρεσία, συγγνώμη, εξωτερικής να αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική Θέλουμε να υπάρξουν ετήσιες εκθέσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι θα υπέρ οι νόμοι που υφίστανται στον τομέα της ανακύκλωσης, για παράδειγμα, όσον αφορά τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, να εφαρμοστούν. Τρίτον, ε, στην έκθεση αυτή ασχολούμεθα με την εξωτερική διάσταση της πολιτικής και της πρώτες ύλε. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει προς τα έξω να αναπτύξουμε μια αξιόπιστη στρατηγική συνεργασίας τόσο έναντι των ε, ε, φτωχών σε πόρους ε, χώρες στην Αφρική για παράδειγμα όσο και έναντι των πλούσιων ε, σε πόρους ε, χώρες, ε, χωρών. στην Ευρώπη οι εισαγωγέ ανακεφαλή είναι περισσότερες σε πρώτες ύλες, είναι περισσότερες από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη γωνιά του πλανήτη. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε μια ευθύνη γιατί σε επενδύσεις για παράδειγμα όσον αφορά την εκμετάλλευση των αποθεμάτων σε τρίτες χώρες θα πρέπει η ΕΤΕ και η Επιτροπή να εξετάσουν κατά πόσο μπορούν να ενταχθούν στις δραστηριότητες σε μια στρατηγική κατά τις φτώχειας. Δηλαδή να θεσπιστούν κάποιοι νόμοι όσον αφορά την ε, διαφάνεια όπως το Frank Act ε, στην Αμερική ή το Publish What You Pay, αυτή η βασική αρχή. Ε, θα πρέπει δηλαδή να μην εξυπηρετήσει η πολιτική μας ε, τα δικά μας συμφέροντα αλλά να τθεί στην υπηρεσία των συμφερόντων και των φτωχών χωρών. Είμαι σίγουρη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σε πολλά διεθνή όργανα να συμβάλλει σε μια διεθνή διακυβέρνηση για τις πρώτες ύλες Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπιτικόφερ και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο κύριο Ταζάνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα αρχίζοντας την ομιλία μου να ευχαριστήσω επισήμως ε, τον εισηγητή, τον κύριο Μπιτικόφερ, για την έκθεσή του. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλες και όλους όσους ε, βοήθησαν ε, τον εισηγητή για την ε, εκπόνηση αυτής της έκθεσης, διότι πρόκειται για μια εξαιρετικά επικοδομητική έκθεση, κατά τη γνώμη μου. Εξάλλου ακολουθεί την, τον ίδιο προσανατολισμό που έχει επιλέξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να προσεγγίσει με στρατηγικό τρόπο αυτό το τόσο κέριο θέμα των πρώτων υλών. Ε, γι' αυτό και επίστηνα από την έκθεσή σας, ε, ε, το επαναλαμβάνω, ότι συμφωνεί το πνεύμα που διέπει την έκθεσή σας πλήρως με το πνεύμα που διέπει τις εργασίες και τους προσανατολισμούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, εξετάζεται όλα τα προβλήματα από όλες τις πιθανές οπτικές ε, γωνίες και εξετάζεται και τις ε, μελλοντικέ κινήσεις μας και τις διάφορες εναλλακτικές πολιτικές λύσεις. Κατόπιν κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες συστάσεις μέσα στην έκθεσή σας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι με τις προτάσεις που κάνετε αναβαθμίζετε τη στρατηγική που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου έχει καθοριστική σημασία. Εδώ και μήνες συνεργαζόμαστε με τον κύριο Μπιτικόφερα μόνο, ε, για αυτό το θέμα των πρώτων υλών. ο κύριος Μέρκης, ο κύριος ε, φέρε διάφοροι βουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Ο στόχος μας, μεταξύ των στόχων μας, είναι να ιδρύσουμε ένα δίκτυο μέχρι το 2012 για τις σπάνιες υγιές και ελπίζω ε, να συμβάλλω και εγώ ούτως ώστε να εγκαταστήσουμε μια πραγματική, μια ουσιαστική εταιρική σχέση για τις πρώτες ύλες. Σε επίπεδο πολιτικής είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το αναφέρατε και εσείς κύριε Βιωτικόφερ στην έκθεσή σας. Εγώ στο ταξίδι από το Μόναχο μέχρι το Στρασβούργο διάβασα προσεκτικά την έκθεσή σας και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ε, το εξής απόσπασμα. Εκεί ε, λέτε ότι η απόκτηση των πρώτων υλών ε, αρχίζει να αποκτά πλέον στρατηγική σημασία. Και ο κ. Μπιτικόφερ αναφέρει στην έκθεσή του ότι το ποσοστό που στην παραγωγή που αφιερώνονται στις πρώτες ύλες ε, υπερβαίνει το ποσοστό που διοχετεύεται στο εργατικό δυναμικό. Αυτό με καταπλήσει. Μιλάτε για μια πιο αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών μέσω της ανακύκλωσης, και τα λοιπά. Βεβαίως, όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία συναποτελούν τη στρατηγική μας και συμφωνούμε. Κατόπιν, το θέμα καινοτομία ε, είναι απαραίτητο αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε τη στρατηγική των πρώτων υλών της Ένωσης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλους τους κρίκους αλυσίδας, δηλαδή από την έρευνα, την εξόρυξη, τη μεταποίηση, την ανακύκλωση ε, θα πρέπει λοιπόν να ε, δημιουργήσουμε μια νέα εταιρική σχέση για τις πρώτες ε, ύλες. Είναι απαραίτητο αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Ο κύριος Μπιτικόφερ είναι αισιόδοξο. Φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς κάποιων κρατών μελών, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι πια παρελθόν διότι το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας έχει δώσει ήδη το πράσινο φως. Ε, το σημαντικό τώρα είναι να ε, αποφασίζουμε με ποιο τρόπο θα υλοποιήσουμε αυτή την εταιρική σχέση. Ένα άλλο σημείο στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς κύριε Μπιτικόφε που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η διπλωματία των πρώτων υλών. Σε όλες τις διεθνείς σχέσεις μας πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη αυτό το θέμα. Είτε πρόκειται για εμπορικέ σχέσεις είτε όχι. Με τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία εξάλλου έχουμε ήδη σημειώσει πρόοδο και έχουμε ε, μια στενότερη συνεργασία σε σχέση με το παρελθόν. Με την Αφρικανική Ένωση έχουμε επίση κοινό σχέδιο δράση ε, και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκής Ένωση υπάρχει κοινή βούληση συνεργασία για το θέμα των πρώτων υλών, λαμβάνοντας υπόψη τι δυνατότητε που έχει ε, η Αφρικανική Ήπειρο σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο ε, Ήπειρου, σε επίπεδο περιφέρεια, περιοχή ή σε επίπεδο χώρας. Ε, ίσως σε μια διάσκεψη για τις πρώτες ύλες θα μπορούσαμε να συμμετήσουμε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για τις πρώτες ύλες ε, τώρα να, να σας πω ότι ε, ε, έχω ταξιδέψει στη Μόσχα, στην Κίνα. Τέλος πάντων εργάζομαι σε πολλά μέτωπα για το ίδιο θέμα. Υπογράψαμε και μία συμφωνία με την Χιλή και ενδέχεται με την Αργεντινή και τη Βραζιλία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να υπογράψουμε επίσης συμφωνία και μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για, για τους βασικούς παραγωγούς λιθίου που έχει τόσο μεγάλη σημασία στον τομέα των ε, πρώτων υλών. Πάντως, ε, όλοι δείχνουν ενθουσιασμό ε, για αυτή την νέα εταιρική σχέση ε, οι πρόεδροι αυτών των χωρών έχουν αναλάβει ε, ούτως ή άλλως δέσμευση για αυτό το ζήτημα. Σχετικά τώρα με τον, ε, τη το βιώσιμο χαρακτήρα της πολιτικής μας, οφείλουμε να επιμείνουμε ώστε να γίνονται σεβαστά τα περιβαλλοντικά πρότυπα κατά την εξόρυξη των πρώτων υλών. Χρειαζόμαστε ως εκ τούτου και την έρευνα και την καινοτομία για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Πάντως ε, θα έπρεπε ε, να διερωτηθούμε πώς ε, θα εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στις σπάνιες γης. Πρέπει να ρωτηθούμε πώς θα εξορίσονται αυτά τα ε, με τα λεύματα και θα συνεργαστώ με τον Επίτροπο Ποτόσνικ ε, στενά. Πρόκειται για μεικτή αρμοδιότητα Ένωση και κρατών μελών. Ε, έχουμε πλήρη επίγνωση. Εμεί θα λειτουργήσουμε ω καταλήτη. Υπενθυμίζω ότι η αρμοδιότητα είναι βασικά των κρατών μελών. Επίση, υιοθετήσαμε την περασμένη εβδομάδα μια βασική εμβληματική πρωτοβουλία για αυτά τα στοιχεία και δίνονται συγκεκριμένε απαντήσει. Πρόκειται για το θέμα τη ανακύκλωση, όπω γνωρίζετε και θα ήθελα να προσθέσω ότι συνεργάζομαι στενά και με την κυβέρνηση της ε, Σουηδίας. Ε, πριν από τις ε, καλοκαιρινές διακοπές έγινε μια πάρα πολύ σημαντική συνεδρίαση για τις δυνατότητες εξόριξης στη θάλασσα του Μπαρένς και μετέβη στη Σουηδία και συνεργάστηκα με τους υπουργούς ε, γι' αυτό το θέμα. Επίσης ε, θα πάω και στην Γρυλανδία όπου θα συζητήσω με τον Πρωθυπουργό της χώρας ε, για το ίδιο θέμα. Η Γρυλανδία διάγεται θετικά ως προς μια μακροπρόθεσμη κοινή στρατηγική σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πρώτες ύλες. Αυτά κάνουμε. Ζητώ συγγνώμη αν ε, μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι αξίζει λόγω της, ε, του ειδικού βάρους ε, που έχει αυτό το ζήτημα. Οφείλουμε να είμαστε διεξοδικοί όταν το εξετάζουμε. και επίσης κλείνοντας να πω ότι προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και ευελπιστώ ότι θα έχουμε τις απαιτούμενες απαντήσεις για τη βιομηχανία χωρίς όμως παρόλα αυτά να πλήξουμε το περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε Ταγιάννη. Τώρα ο κύριος Μπρόκ είναι στο, ο πρώτος ομιλητής, αλλά δεν τον βλέπω, οπότε θα ακούσουμε την κυρία Σνίμπερ Γιάστραμ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν ως ήθιστε εδώ στο Κοινοβούλιο να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μπιούτι για αυτή την έκθεση. Ως ε, εισηγήτρια ε, για πολιτική υπέρ της ανάπτυξης. Είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων προς την Ήτρε γιατί πραγματικά συμπέλευε πολλά ρεθίσματα από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Όπως είπε ο κ. Μπιουτικόφερ, ε, όσον αφορά τις πρώτες ύλες, εδώ πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι μείζονος σημασίας. Μέχρι το 2050 υπολογίζουν τα Ηνωμένα Έθνη μία αύξηση της τάξης του 300% όσον αφορά την ζήτηση των πρώτων υλών. Και ιδιαίτερα σημαντική είναι αυτή η συζήτηση επίσης σε σχέση με, ένα, μια συνεκτική πολιτική ανάπτυξης. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω ένα παράδειγμα. Εναπτυσσόμενες χώρες χάνουν ε, ε, λόγω κακών ε, πραγμα... Ε, κακών πρακτικών και λοιπόν ε, συμφωνιών ετήσια 80 έως 160 τρισεκατομμύρια δολάρια και αν δούμε ποια είναι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ είναι 8-3 ε, το χρόνο. Δηλαδή αυτό το οποίο εμείς ε, δίνουμε σε σχέση με αυτό το τεράστιο νούμερο είναι σταγόνα στον ωκεανό. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό ε, ότι η έκθεση επισημαίνει τις πρωτοβουλίες διαφάνειας όπως το ATE και θα πρέπει οι πρωτοβουλίες αυτές να είναι μακροπρόθεσμες και θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις εκ μέρους του Joint Africa Action Plan όσον αφορά για παράδειγμα τη διαπραγμάτευση κάποιων συμφωνιών με εταιρείε πρώτων υλών. Κάθε ευρώ το οποίο χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς ε, κομίζει στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες μια υπεραξία των 10 ευρώ και μπορούμε να πούμε δικαιολογημένα ότι συνιστά αποτελεσματική μορφή βοήθειας σε αντίθεση με κάποια άλλα μπαλώματα εκ των υστέρων. Ευχαριστούμε πολύ ε, κυρία Σνίμπερ. Ο κύριος ε, Λάγκε. Παρίστατε, παρίστατε. Έχετε το λόγο κύριε Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Σιγητά και από τη δική μου πλευρά ε, ευχαριστούμε πολύ για την ιδιαίτερως απαντητική αυτή έκθεση και τη σημαντική εργασία που επιτελέσατε. Κύριε Επίτροπε, η πολιτική των πρώτων υλών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Και επίσης η διάσταση του εμπορίου είναι ιδιαίτερα καθοριστική και υπό την έννοια αυτή θεωρώ ότι είναι ορθό και δικαιολογημένο η πολιτική των πρώτων υλών ε, στο διεθνές πλαίσιο να διαμορφώνεται υπό το πρίσμα της βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρώπη. Και ε, εδώ νομίζω τα επιμέρους σημεία είναι καθοριστικά. Ε, νομίζω ότι εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε τις πρώτες ύλες στον κόσμο μέσω σύναψης εταιρικών συμφωνιών, ε, μπορούμε να το πράξουμε μόνο εφόσον οι εταιρείε Ε, των πρώτων υλών ε, συμπεριφέρονται σωστά. Δεν είναι δυνατό να φοροδιαφεύγουν οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίε ή να βάζουν τους ανθρώπου να εργάζονται υπό αναξιοπρεπεί συνθήκε. Γι' αυτό, εάν θέλουμε να κερδίσουμε πρώτε ύλε, θα πρέπει οι επιχειρηματίε να τηρούν ξεκάθαρε κοινωνικέ και περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτες ύλε οι οποίε χρησιμοποιούμε να μην προέρχονται από περιοχέ, από ζώνε κρίσεων ε, και να μην χρηματοδοτούνται από ομάδες που θέλουν να κερδίσουν χρήματα από αυτό και να κάνουν φίλους πολέμους. Χρειαζόμαστε ένα διεθνές σύστημα χρηματοδότησης για την άντληση των πρώτων υλών και για τις εμπορικές αλυσίδες, ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε από πού προέρχονται. Άλλωστε υπάρχουν καλά αποτυπώματα της πρώτης ύλες παντού. Τρίτον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να μην ε, γίνεται, γίνονται παράνομες εξαγωγές των πρώτων υλών ε, θα πρέπει να δούμε τις τρύπε στην νομοθεσία Καρλ Χάιντς Φλόρεντς αλλά θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τους ελέγχους όταν για παράδειγμα σε ένα ευρωπαϊκό λιμάνι μόνο ένα άτομο θα πρέπει να εξασφαλίσει όλο τον έλεγχο σίγουρα δεν είναι επαρκής. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να ελέγχουμε καλύτερα τις εξαγωγές και να εξασφαλίσουμε οι μονοπελιακές και ολιγοπολιακές δομές στο εμπόριο των πρώτων υλών να καταργηθούν. Και εδώ, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή κάνει τα σωστά βήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπιουτικόφερ και κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάγκε. Η κυρία Μέρκης έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Σιγητά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το έγγραφο αλλά και για τη στρατηγική και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους ε, που έχουν συνεισφέρει μέχρι τώρα στη συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα αποφέλης και μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα ε, προς τα εμπρός. Πρέπει να ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να προλάβουμε μία επόμενη κρίση αν εκινήσει η ανάπτυξη. Σίγουρα χρειάζονται πρώτες ύλε, ε, θα είναι μεγάλες οι ανάγκες ε, και ίσως αν δεν υπάρχουν να υπάρχει μεγάλη πίεση στην δεχόμενη μελλοντική ανάκαμψη. Έχει αδυναμίες η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό και θα πρέπει να δούμε πώς εντός ε, της Ένωσης θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα απόβλητα. Σε ό,τι αφορά τις πρώτες θα πρέπει να υπάρξει ανακύκλωση και βέβαια η καινοτομία πρέπει να ευνοηθεί, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη αποκρισταλωθεί ιδιαίτερα. Θα πρέπει να δούμε επίσης τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά όχι μόνο, πώς θα μειώσουμε την εξάρτηση που έχουμε σε διάφορους τομείς. Θα πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορές, οι θα πρέπει οι πολίτε αλλά και η βιομηχανία να αλλάξει. Χρειαζόμαστε ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Γίνεται λόγο ε, για την διακυβέρνηση, για τις τράπεζε. Δεν μιλάω για κάτι αντίστοιχο όμω, μιλάω για βαθιές αλλαγές, για τομέ στην οικονομία. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, θα πρέπει να γίνουν ε, προσπάθειες ε, προς την πρόθεση καλύτερων ποιοτικά αλλά και φιλοπεριβαλλοντικότερων προϊόντων. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, ε, πάση θυσία, είναι να προστατεύσουμε και να σεβαστούμε τη φύση. Γιατί πολλές φορές κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε αυτή την πτυχή του προβλήματος. Μήπως οι πόλεις ε, κάθονται πάνω σε πραγματικά χρυσορυχεία, σε κοιτάσματα, τα οποία θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα, να τα αξιοποιήσουμε περισσότερο. Δεν θα πρέπει να δούμε και αυτό το ζήτημα. Οι συνάδελφοί μου έχουν διατυπώσει πολύ καλές προτάσεις. Και ελπίζω να καταφέρουμε να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές και να δείξουμε όλη την απαιτούμενη υπευθυνότητα. και καινοτομία. Είναι κάτι που πραγματικά θεωρώ πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάρμπου είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Σεγητά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις πρώτες ύλε, αλλά και την πρόταση εκπόνησης μιας στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι τα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να τέχουν ιδιαίτερη ε, προσοχή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την ανάγκη να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντιμετωπίζουμε πολλέ προκλήσει ό,τι αφορά τι πρώτε ύλε στη γεωργία. Επίση, πολλέ φορέ γίνεται λόγο για τι διακοιμάσεις ε, των τιμών στι αγορέ ή μιλάμε για την ε, μείωση των τροφίμων, μιλάμε για τις λειτουργίες ε, στην ε, τροφική αλυσίδα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η στρατηγική που θέλουμε να εκπονήσουμε θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους φραγμούς στις εξαγωγές, τα εμπόδια στις εξαγωγές. Το κείμενο δεν είναι ιδιαίτερα σαφές σε ό,τι αφορά αυτή την πτυχή, την πτυχή του ΠΟΕ. Θα πρέπει να διασαφινιστούν αυτές οι πτυχές και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των γεωργικών αγορών και γεωργικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό η στρατηγική θα είναι αποτελεσματική και θα εξασφαλίσει και την ασφάλεια του εφαντισμού σε τρόφιμα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στους ομιλητές ε, των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Κυρία Ντελκαστήγιο είναι η πρώτη ομιλήτρια, μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε μια έκθεση την οποία έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούσε τότε τη στρατηγική για την αντιμετώπιση ενός πολύ σημαντικού ζητήματος που δεν είναι άλλο από τη διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών και την αύξηση της ζήτησης πρώτων υλών από τις αναπτυσσόμενες χώρες και όλες ιδιαίτερως από την Κίνα. Η δική μου πολιτική ομάδα θα ήθελε να πει ότι συμφωνεί επί της ουσίας με την έκθεση Μπουτικόφερ γιατί θεωρούμε ότι κάνει μια προσέγγιση και δίνει μια ε, εστίαση πάρα πολύ ικανοποιητική στις πρώτες ύλες και στη στρατηγική για την χρήση, την πρόσβαση και την ανάπτυξη από τον υλών. Νομίζουμε ότι υπάρχει ισορροπία στην έκθεση, την έκθεση την οποία συζητούμε σήμερα. Ισορροπία μεταξύ της πρόσβασης στις πρώτες ύλες που είναι πάρα πολύ σημαντικές και απαραίτητες και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπογραμμίζεται σωστά η ανάγκη να χρησιμοποιούνται σωστά οι πηγές πρώτων υλών και επίσης η έκθεση διατυπώνει μια σειρά προτάσεων που είναι πάρα πολύ απαραίτητες για να βελτιωθούν οι πρακτικές της ανακύκλωσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όνομα τη πολιτική μου ομάδα θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα πρέπει το θέμα αυτό να το προσεγγίσουμε όχι μόνο από, όχι από την πλευρά τη μείωση τη κατανάλωση, γιατί ε, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να διατηρηθεί και πρέπει να τονωθεί, να ενισχυθεί. Αυτό που πρέπει λοιπόν να προτείνουμε είναι πολιτικέ αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών και πολιτικέ οι οποίε πραγματικά δίνουν κίνητρα, παρακινούν προς ε, τη να τη χρήση αυτών των πρώτων υλών. Επίσης, ε, αυτό θα επηρεάσει θετικά και τις κερδοσκοπικές ε, πρακτικές, γιατί νομίζω ότι οι προτάσεις της Κομισιόν θα οδηγήσουν στο να έχουμε μια πιο διαφανή αγορά σε σχέση με το πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Άρα μια αγορά όπου οι δυνατότητες κερδοσκοπίας θα είναι μικρότερες. Η κυρία Ούλσκοκ, τώρα από πλευρά των σοσιαλιστών έχετε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους Γιούντιτ Μάρκης, κύριο και με τον εισηγητή τον κύριο κόφερ. Ήδη είπαν τα σημαντικά, δηλαδή πιο αποτελεσματική χρήση των ε, πρώτων υλών, ε, η ανάκτηση των σπάνιων γεών από τα απόβλητα, η ανακύκλωση, μόνο αυτά μπορούν να εξασφαλίσουν προστασία του περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε καινοτόμια, χρειαζόμαστε νέες τεχνολογίες, μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Θα ήθελα όμως εγώ να τονίσω μια τελώς διαφορετική διάσταση ε, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους ψηφοφόρους μου. Ε, το Κοινοβούλιο ε, ασχολήθηκε ε, με το θέμα των πρώτων υλών στον όταν στη Βόρεια Σουηδία. Πήγανε οι ειδικοί του Κοινοβουλίου στη Βόρεια Σουηδία για να δουν τι σημαίνει η εξόριξη αυτών των σπάνιων γεών. Πήγα λοιπόν και συνάντησα με εκπροσώπους της βιομηχανίας, με συνδικαλιστικές οργανώσεις, με όλους τους ενδιαφερομένους και μου είπαν ότι αυτός ο παλιός ε, τομέας, αν θέλετε, πλουτοπαραγωγικός πόρος ε, αποκτά μια νέα λάμψη και τώρα ε, προσπαθούμε να βρούμε νέες τεχνικές για να αναβαθμίσουμε την εξόριξη λόγω της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης για αυτές τις πρώτες ύλες. Η παγκοσμιοποίηση ουσιαστικά μας τρέφει πίσω στην Ευρώπη, ενώ αρχικά είχαμε εστιάσει την προσοχή είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι πάρα πολύ συναρπαστικό αυτό το θέμα και θα ήθελα να πω στον ε, Επίτροπο ε, ότι δεν χρειάζεται να πάμε στη Γρυλανδία. Έχουμε ολόκληρη Βόρεια Ευρώπη εδώ. Έχουμε πάρα πολλά πάρα πολύ υψηλή ε, τεχνογνωσία, έχουμε καλές συνθήκες εργασίας, έχουμε σπάνιες πρώτες ύλες ε, ε, και οι αξιοπρεπές συνθήκες εργασίας έχουν μεγαλύτερη σημασία γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στον τομέα της εξόρεξης. Και δεν χρειάζεται να στρέφουμε το βλέμμα μας μακριά από την Ευρώπη, στη Γρυλανδία. Έχουμε εδώ αυτά που μας χρειάζονται. Η πολιτική των πρώτων, για τις πρώτες ύλες επίσης, έχει ε, αποφασιστική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βόρεια Ευρώπη έχει καθοριστικό ρόλο για την βιομηχανική ανάπτυξη. Αυτό ήταν ένα βασικό μήνυμα από την επίσκεψή μας στη Βόρεια Σουηδία. Εκεί υπάρχουν και υποδομές ε, και για τα βιομηχανικά κέντρα και για την εξόρυξη των πρώτων υλών. Και όλα αυτά έχουν κέρια σημασία για τη μελλοντική βιομηχανική ανάπτυξη. Με αυτή την έκθεση ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκριθούν νέες κατευθύνσεις γραμμές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, και οι κατευθυντήριες γραμμές ε, που υπάρχουν ε, βάσει του ερευνητικού προγράμματος πλαισίου να εφαρμοστούν στις εξωτερικές βιομηχανίες. Πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να καταθέσει σχετικές προτάσεις. Και κάτι άλλο που ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι είναι σχετίζεται με την εξόριξη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται αυτή η εταιρική σχέση από ισότητα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε ε, να επιστρέψουμε στην ε, παλιά εποχή της απικιοκρατίας. Ε, δεν μπορούμε να περιέλθουμε πάλι σε αυτή την ετεροβαρή σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει να προωθήσουμε μια ισότιμη εταιρική σχέση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ δούμε. Η κυρία Εκ τώρα από πλευρά ε, των φιλελευθέρων για τρία λεπτά. Ε, Ευχαριστώ. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία από τις βασικότερες προκλήσεις σήμερα. Οι Ευρωπαίοι ζουν μέσα σε ένα όλο ένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Έχουμε νέες προκλήσεις ε, για να εξασφαλίσουμε ε, την οικονομική ευρωστία και να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να αναδιαρθρώσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία για να έχουμε την ευφύ, βιώσιμη και ισότιμη ανάπτυξη για όλους. Αυτές είναι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μέσα στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και επίσης ε, θα πρέπει να είναι αυτό το χαρακτηριστικό της μελλοντική πολιτικής μας για τις πρώτες ύλες. Μην υποτιμάτε αυτές τις προκλήσεις βάσει κάποιων εκτιμήσεων. Χρειάζονται επενδύσεις για τις μεταφορές, για την ενέργεια, για τις, ε, ε του ύψου ε, των 4.000 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2020 και οι πρώτες ύλες είναι το κλειδί για τις μελλοντικές επενδύσεις μας αν θέλουμε να έχουμε ηγετικό ρόλο. Ε, επίσης όσο πρασινοποιούνται οι οικονομίες τόσο ανταγωνίζονται βασικά για τις πρώτες ύλες ε, που όμως εισάγουμε εμείς από ανταγωνιστικές δυνάμεις ε, μέχρι στιγμής. Επίσης πρέπει να συνδέσουμε την πολιτική για τις πρώτες ύλες με άλλες πολιτικές, τη βιομηχανία, την έρευνα, το εμπόριο, τις μεταφορές, τη βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό διότι για να αντιμετωπίσουμε την κρίση χρειαζόμαστε πραγματι... μεταρρυθμίσεις ε, που να εστιάζονται, να στρέφονται προς τη μελλοντική ανάπτυξη. Η πολιτική των πρώτων υλών πρέπει να συνδυαστεί λοιπόν με άλλε πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στι πρώτε ύλε ε, για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Ε, ε, πέρα η πολιτική για τι πρώτε ύλε Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από το να είναι πράσινη και να προσανατολίζεται προ την ανάπτυξη, πρέπει να φροντίζει ώστε να έχουμε μια ισότιμη σχέση με αυτού που μα παρέχουν τι πρώτε ύλε. Οι τρίτε χώρε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον αναπτυξιακό μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, κυρίω σε χώρε που εξέρχονται από μια ένοπλη σύραξη, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν οι πρώτε ύλε για να χρηματοδοτήσουν σειράξει ή για την περαιτέρω κλιμάκωσή του. Ε, Επίση, ε, κατάργηση των εμπορικών φραγμών ε, στι τρίτε χώρε. Αυτή πρέπει να είναι η πολιτική μα και όχι να αποθεματοποιούμε εμεί τι πρώτε ύλε υπονομεύοντα τη δημοκρατία σε αυτέ τι χώρε. Επίση πρέπει να αξιοποιήσουμε τι πρώτε ύλε που έχουμε ήδη στην Ένωση. Συχνά διστάζουμε, αλλά ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαρκή σε πόρου. Έχουμε πετρώματα, έχουμε δάση. Κυρίω η Βόρεια Ευρώπη έχει το απαιτούμενο δυναμικό για να μα δώσει με βιώσιμο τρόπο τι πρώτε ύλε που χρειαζόμαστε ε, και με, τον στρατη... με τη στρατηγική διαχείριση των δικών μας επόνων ε, σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση της εσωτερικής αγοράς θα μπορέσουμε να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αυριανή οικονομία και κλείνω ε, συγχαίροντας τον εισηγήτη. Thank you, Madam Mr. on behalf of the... Κύριος τώρα έχει το λόγο από πλευρά των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε εισηγητά. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο εισηγητή ε, και τον κύριο Ταγιάννη για τα όσα είπε ε, φαίνεται υπάρχει συμφωνία. Όλοι επιθυμούν μια σωστή στρατηγική για τι πρώτε ύλε, αλλά θα πρέπει κάπω να οξύνω του τόνου. Διαβάζοντα αυτή την έκθεση και την έκθεση τη Επιτροπή, διαπιστώνω ότι υπάρχουν τεράστιε διαφορέ και χαίρομαι πολύ που ο κύριο Ταγιάννη χαίρεται για την έκθεση του Κοινοβουλίου. Αλλά τελικά η στρατηγική θα είναι διαφορετική, γιατί στην έκθεση τη Επιτροπή ε, το θέμα είναι ο αγώνα με την Κίνα για τι ε, διεθνεί πρώτε ύλε που θα πρέπει να έρθουν στην Ευρώπη. Ευρώπη. Ε, ε, νομίζω ότι είναι σφαλμένη ε, σειρά πραγμάτων. Θα πρέπει να είμαστε αποδοτικοί με τους δικούς μας, με τις δικές μας πρώτες ύλες. Ένα απλό παράδειγμα, η ανακύκλωση. Εάν έχουμε, για παράδειγμα, ένα τόνο σε ένα ορυχείο και βρούμε εκεί δύο γραμμάρια, μπορούμε να βρούμε δύο γραμμάρια χρυσό. Ε, σε απόβλητα κινητών μπορούμε να βρούμε 150 γραμμάρια χρυσού. Ε, αυτό είναι πολύ φτηνότερο. Ε, νομίζω λοιπόν κύριε Επίτροπε ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε στην ανακύκλωση των δικών μας πρώτων υλών και τα ορυχεία να μην τα φτιάξετε στι ε, περιοχέ Natura 2000. Αυτό το αναφέρει η έκθεση. Λέτε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον, αυτό θα πρέπει να γίνει ε, ξεκάθαρο, όχι σε περιοχέ τη Natura 2000 και όχι στον Βόρειο Πόλο. Γιατί ε, και εκεί θα πρέπει να κρατηθεί απ' έξω η Ευρώπη. Άρα πρόκειται για μια συγκεκριμένη χάραξη πολιτική και όχι για μεγάλο λόγια. Και τρίτον, όταν πάμε εκτός της Ευρώπης στην επαφή με τις αναπτυσσόμενες χώρες, εδώ το ζητούμενο είναι η διπλωματία. Αλλά αυτό πρέπει να περάσει από όλη την ε, Επιτροπή και από τον Επίτροπο Εμπειρίου, Και εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το λόγο έχει η κυρία Γκέρλινγκ, εξ μέρους των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επίση να εκφράσω τι ευχαριστίε μου για τον εισηγητή για την έκθεση που διάβασα μεγάλο ενδιαφέρον. Ακολούθησα την έκθεση αυτή ω σκιώδη εισηγήτρια στην Επιτροπή Περιβάλλοντο και η συζήτηση εκεί επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένου τομεί τη έκθεση. Είναι απολύτω ξεκάθαρο θα πρέπει να εξετάσουμε κάποιε στρατηγικέ για τη μείωση για την ε, αύξηση της ανακύκλωσης των πρώτων υλών. Αλλά δεν θα πρέπει να περιπλέξουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Η στρατηγική είναι μια στρατηγική. Ο τίτλο τη εισήγηση είναι αποτελεσματική στρατηγική. Ε, θα πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι ίσω είμαστε υπερβολικά περιγραφικοί και συγκεκριμένοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε ένα περιθώριο. Για παράδειγμα, ε, την αστική εξόριξη, το urban mining. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου υπάρχει μια μακρά ιστορία χωματων ε, ε, και νομίζω ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί δημιουργούνται εκπομπές αερίων θερμοκηπίων μέσω των χωματιρών και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Επίσης ε, μπορούν ε, να δημιουργήσουν τοξικά αέρια, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν συνεχίσουμε με αυτή, στη βάση αυτής της στρατηγικής και θα πρέπει να έχουμε πολύ προσεκτικές μελέτες επιπτώσεων περιβάλλοντος. Ε, ε, πολλή συζήτηση γίνεται για ε, θέματα διαστρέβλωσης αγοράς και χειραγώγηση της αγοράς και κερδοσκοπίας. Όλα αυτά είναι ανοιχτά προς συζήτηση, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο που θα πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να συζητάμε για αποθεματοποίηση, γιατί αυτό ισοδυναμεί με μια χειραγώγηση των αγορών και νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα μας πάει παραπέρα. Χαιρετίζω λοιπόν την έκθεση. Όπως είπα, ευχαριστώ τον εισηγητή και αναμένω με ανυπόμονα την ε, συνεργασία για την εκπόνηση της στρατηγικής για τις πρώτες ύλες, γιατί έχουμε ένα μακρό δρόμο να διαρνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέρλινγκ. Τώρα ο κύριος Ματίας εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ αρχίζοντας να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε την περιγραφή των τωρινών αναγκών της βιομηχανίας ως προς τις ε, πρώτες ε, ύλες. Ε, και την ε, έμφαση για τους περιβαλλοντικούς ε, κινδύνους και τα όσα λέει για την πολιτική της ανακύκλωσης. Όλα αυτά είναι θετικά επιμέρους στοιχεία της έκθεσης και σας συγχαίρω. Θα ήθελα όμως να σχολιάσω εδώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να συμφωνήσω με αυτή την επωνομαζόμενη διπλωματία των πρώτων υλών. Αυτή η πρόταση σε συνδυασμό με την πρόταση θέσπισης ενός συστήματος εποπτείας σε επίπεδο G8 ή G20 ουσιαστικά διευρύνουν κατά τη γνώμη μου ε, μια παλιά διχοτόμηση του κόσμου, δηλαδή ανάμεσα στις βιομηχανικές χώρες με πολύ αυξημένες ανάγκες ω προς τις πρώτες ύλες και θεμητές ανάγκες έτσι και αφετέρου ε, τις ε, φτωχές χώρες που είναι πλούσιες όμως σε πρώτες ύλες πλην όμως δεν μπορούν να τις εκμεταλλευτούν. Ξέρουμε ότι η βάσει της τωρινής βιομηχανικής συγκυρίας υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να προωθήσουν την πάση θυσία εκμετάλλευση των πρώτων Όμω Όμως πρέπει να αλλάξουμε σε σχέση με το παρελθόν. Ας κοιτάξουμε τι έγινε με τα 15 χρόνια, ε, με τα, ε, συγγνώμη, τους πέντε τελευταίους αιώνες ε, της εκμετάλλευσης τη Ευρώπης από πλευρά της Ευρώπης αυτών των χωρών. Αυτές οι χώρες δικαιούνται ισότιμη μεταχείριση κατά την εκμετάλλευση των ε, πρώτων υλών του ε, και νομίζω ότι η υπηρεσία εξωτερική ε, δράση θα πρέπει να αποσκοπεί στη συνεργασία και όχι στη διπλωματία των πρώτων υλών. Πασκά. Ευχαριστούμε, Παμπασκά. Από την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, όπως ε, αναφέρεται στην έκθεση του κυρίου Βιδικόφερε, η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει αυξανόμενες δυσκολίες ε, για να βρει τους απαιτούμε, τις απαιτούμενες πρώτες ύλες ε, για ταχεία οικονομική ανάπτυξη, βιομηχανική ανάπτυξη. Ε, επίσης, από πλευράς ε, ε, Αμερικής αυξάνεται η ζήτηση των σπάνιων γεών και έτσι αυξάνονται οι τιμές σε ολόκληρο τον κόσμο και πιέζεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όμως πολλά βιομηχανικά προϊόντα που θεωρούνται απόβλητα εμπεριέχουν τέτοια σπάνια μέταλλα και άλλες τέτοιες ουσίες που συχνά εισάγουμε από το εξωτερικό εμπορική διπλωματία είναι ένας ε, τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην ανακύκλωση ε, των πρώτων υλών. Ε, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι πηγή μόλυνσης, είναι τρόπος απόκτησης πόρων πρώτων υλών για να μην εξαρτώμεθα από τις χώρες που εξάγουν αυτές τις πρώτες ύλες. Ο κ. παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκβαση της συζήτησης σχετικά με τη στρατηγική της ευρωπαϊκής ένωσης για τις πρώτες ύλες αλλά και για την υψηλή ποιότητα της τελικής έκθεσης που τίθεται σε ψηφοφορία ενώπιον της ολομέλειας. πιστεύω ότι το τελικό κείμενο εμπεριέχει πραγματικά εκείνες τις παραμέτρους αναπτυξιακές βιομηχανικές περιβαλλοντολογικές και ανατομικές που οφείλουν να διέπουν μια δυναμική ευρωπαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρώτες ύλε. Ζητούμενο είναι μια στρατηγική η οποία θα ενισχύει τις αναπτυξιακές δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα στηρίζει αλλά και θα στηρίζεται από την ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή. Θα αξιοποιεί τις εγχώριες πρώτες ύλες υπό συνθήκες απολύτου σεβασμού του περιβάλλοντος θα συνδέεται με την ερευνητική και καινοτομική προσπάθεια με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία και την εκπαίδευση υψηλή ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού. θα ισχυροποιεί τη θέση τη ευρωπαϊκή ένωση μέσα σε ένα ευμετάβλητο διεθνέ περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμό για την πρόσβαση στου φθήνοντε φυσικού πόρου αναμένεται να είναι όλο και σκληρότερο. κύριε πρόεδρε θα ήθελα να σταθώ στο θέμα των σπανίων υγειών στο οποίο επανειλημμένα έχω αναφερθεί από αυτό το βήμα προσωπικά αισθάνομαι δικαιωμένο για την επιμονή μου στην ανάδειξη αυτού του θέματος και τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την ευρωπαϊκή επιτροπή. οι σπάνιε γέες από παραμελημένο εξωτικό θέμα για λίγους ειδικού κατέληξαν να βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων και σε άρθρα περιοδικών. λειτουργήσαν σαν ένα χρήσιμο σύμβολο αναδεικνύοντα τι στρατηγικέ εξαρτήσεις τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρώτε ύλε και την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη αποφασιστική πολιτική όπου η βιομηχανική, η ερευνητική και η καινοτομική προσπάθεια θα συνεπικουρούνται από ξεκάθαρες και ισορροπημένες διεθνείς σχέσεις. Αισθάνομαι δικαιωμένος και για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την πρότασή μας για δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων σπανίων υγειών, όπως πρόσφατα τουλάχιστον ανακοίνωσε, προκειμένου να υποβοηθήσει τη σταθερότητα των τιμών και την ομαλή τροφοδοσία τη Ευρωπαϊκή Βιομηχανία πράσινης και υψηλής τεχνολογίας. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο next Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γκίρεκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτική των ε, πόρων Πολλές φορές ε, έχει το κίνδυνο των μονοπωλίων, επειδή υπάρχει ανισομερής κατανομή των πόρων και των πρώτων υλών ε, στον πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί με δίκιο τρόπο τους πόρους. Η ενέργεια ε, είναι απαραίτητη για, την, για τους πόρους και είναι και ένα ε, σπαράγοντας αποτελεσματικότητας. Σε ό,τι αφορά την εξόριξη πόρων, θα πρέπει αυτό να είναι ένα θέμα ε, για τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την υδροδότηση, για την τοπική γεωλογία. Έτσι θα γίνει σεβαστική αρχή της επικουρικότητας και θα υπάρξει και οικονομική αποδοτικότητα. Από τη Ρωσία εισάγουμε πολλούς ενεργειακούς πόρους. Η ανακύκλωση όμως έχει τεράστιο δυναμικό. Βέβαια απαιτεί έρευνα, απαιτεί καινοτομία. Η μηχανική των υλικών, το material engineering, η υποκατάσταση δηλαδή ενεργοβόρων από άλλους είναι ε, ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, δηλαδή η μεγαλύτερη χρήση της ξυλίας στις ε, οικοδομές ή η εναλλακτική ε, η χρήση άλλων υλικών αντί των μετάλλων σε μηχανήματα. Υπάρχουν μεταλλεύματα που έχουν ε, ιδιαίτερε ποιότητε, όπω παραδείγματο χάρη οι σπάνιε Και αυτά τα υλικά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ευχαριστούμε πολύ. Τόιρερ, επόμενο ομιλητή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ καταρχήν τον εισηγητή κύριο Μπιούτι Κόφερ για την εξαιρετικά καλή του έκθεση. Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, κύριε Ταγιάννη, σήμερα κάναμε μια ξεκάθαρη χειρονομία, κάνατε μια ξεκάθαρη χειρονομία και γι' αυτό είναι για μας ένα δείγμα ελπίδας. Γιατί στην προηγούμενη στρατηγική της Επιτροπής δεν είχαν εκπληρωθεί οι προσδοκίες μας. Αλλά στην στρατηγική για τις πρώτες ύλε ε, προσδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στον αφορά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια συνεκτική στρατηγική. Χρειαζόμαστε τρει πυλώνε. Την εξασφάλιση των δικών μα πηγών πρώτων υλών. Δεύτερον, την στρατηγική για την ανακύκλωση και την αύξηση τη αποδοτικότητα. Αλλά χρειαζόμαστε επίση και ένα κοινό διάβημα για να οικοδομήσουμε εταιρικέ σχέσει με του βασικού προμηθευτέ πρώτων υλών στον κόσμο. Οι ε, τροπολογίε των φιλελευθέρων επικεντρώνονται στην ενίσχυση του ρόλου των επιστημόνων και τη συμπερίληψή του σε αυτή τη στρατηγική. Γιατί υπάρχουν πολλέ σύγχρονε τεχνικέ, για παράδειγμα όσον αφορά τι πρώτε ύλε στο βυθό της θάλασσας, του ωκεανούς που μπορούν να αξιοποιηθούν, και, αλλά θα πρέπει πρώτα να εξερευνηθούν, ε, να διερευνηθούν. Και εδώ ε, μπορούν οι ευρωπαϊκές ε, χώρες να κάνουν μια προσφορά προς τις τρίτε χώρες. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται την ιδιαίτερη βοήθειά μας. Οι μεγάλοι όμιλοι μπορεί να εξασφαλίσουν τις δικές τους πρώτες ύλε, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται μια κοινή στρατηγική. Γι' αυτό ας κινηθούμε από κοινού να ε, συσπυρώσουμε τις χώρες μέλη για να χαράξουμε μια περιβαλλοντική πολιτική και να πτύξουμε το διεθνές εμπόριο από κοινού με την αναπτυξιακή πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τόιρερ. Η κυρία Φιγερέιδο είναι η επόμενη ομιλήτριά μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνούμε ότι χρειάζεται μια αποτελεσματική στρατηγική για τι πρώτε ύλε. Ε, θα πρέπει να αποφύγουμε τι καταστάσει που αντιμετωπίσαμε το 2007-2008. Πολλέ πρώτε ύλε έφτασαν σε ε, ε, τρομακτικά υψηλέ τιμέ και λόγω κυρίω τη κερδοσκοπία στι αγορέ πρώτων υλών. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να ισχύσουν οι δίκαιε προποθέσει, όπω και στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Υπάρχουν και στην αγορά πρώτων υλών παράγωγα προϊόντα ε, που διαρκούν πολλά χρόνια και λόγω της κερδοσκοπίας ε, καταργείται η πρόσβαση στις πρώτες ύλες ε, ουσιαστικά και να μην αναφερθώ στην έλλειψη διαφάνειας. Χρειάζεται επίσημη ενημέρωση για τα αποθέματα των πρώτων υλών, για τη μεταφορά τους, για να καταλάβουμε πότε και για ποιους λόγους σταματάει ο αφοδιασμός των πρώτων υλών. Επίσης να εκμεταλλευτούμε το γεωλογικό πλούτο της Ευρώπης ε, ακόμη και υποβρυχίως, υποθαλάσσια. Δηλαδή οι υποθαλάσσιοι πόροι της ε, Ένωσης πρέπει να εκμεταλλευτούν. Ναι, μόνο έτσι θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των χωρών, ναι, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν οι πρώτες ύλες. Ε, βεβαίως θα πρέπει να ισχύσουμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες, κυρίως με αφρικανικές χώρες, βεβαίως αποφεύγοντας οποιαδήποτε νέα μορφή απεικιοκρατίας. Χρειάζεται λοιπόν μια εξερθολογισμένη χρήση και ανακύκλωση επίσης των ε, πρώτων υλών στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ε, για να μην ε, χάνουμε τις πρώτες ύλες, για να δημιουργήσουμε δευτερογενείς πηγές, για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του τέλους κύκλου ζωής κάποιων προϊόντων, για να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για τη βιομηχανία. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνυπολογίζει όλες αυτές τις διαστάσεις του ζητήματος για να εκπονήσει μια αποτελεσματική στρατηγική. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπέλντερν, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες είναι πάρα πολύ σημαντική για την ευμερία των Ευρωπαίων πολιτών. Επομένως, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των αγορών πρώτων υλών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσει να υπάρχει σταθερότητα, διαφάνεια και ρύθμιση ω ένα βαθμό των αγορών. Βέβαια, πρέπει να διαρωτηθούμε μέχρι πού φτάνει αυτή η ρύθμιση. Επίση, η ανακύκλωση, η διαφοροποίηση των πόρων είναι σημαντικά θέματα. Η λέξη κλειδί εδώ είναι η λέξη βιωσιμότητα. Οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ε, πρέπει να ακολουθήσουν υπεύθυνε πολιτικέ. Θα πρέπει να είναι σωστέ ε, οι ε, συνθήκες και οι προϋποθέσεις και όταν γίνεται πρόταση για κάποια μεταλλεύματα τα οποία θα προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, πέσουν θύματα αυτών των προτάσεων ε, οι λαοί των περιοχών αυτών. Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συναλλαγές μας με άλλες χώρες και θα πρέπει να είναι ανοιχτό το εμπόριο αλλά σταθερές οι αγορές. Χίμπνερ είναι η επόμενη ομιλητή. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Ταζάνη και επίσης θα ήθελα ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Μπιούτε Κόφερ, ο οποίος ε, πραγματικά συνέταξε μια πολύ καλή έκθεση. Το σημερινό θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Χρειαζόμαστε τους πόρους, όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος. Μιλούμε για μια στρατηγική που θέλουμε να είναι επιτυχημένη και ε, που θα χαράξει μια νέα κατεύθυνση όσον αφορά την χρήση των ε, πόρων. Οι φυσικοί πόροι είναι η βάση ε, κάθε μορφής οικονομίας για την ευρωπαϊκή οικονομία και την παγκόσμια οικονομία και επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε για να εργαστούμε και υπέρ των μελλοντικών γενεών. Όχι μόνο η δική μας ε, γενιά θα πρέπει να, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους σπόρους, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε κάτι και για την επόμενη γενεά η ευρωπαϊκή οικονομία θα πρέπει να αποβεί ανταγωνιστική, να μειώσει τις εκπομπές του του άνθρακα και θα πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με το ζήτημα των αποβλήτων που ε, ε, περιέχουν ε, πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Ε, ο δρόμος αυτός θα, για την παγκόσμια οικονομία θα είναι δαπανηρός, αλλά χρειάζονται και πολλές αλλαγές σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε σύγχρονες τεχνολογίες, χρειαζόμαστε νέες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Η πολιτική μας θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντικό η στρατηγική μας να μην ε, ε, ε, σκέφτεται μόνο τη δική μας γενιά αλλά και τις μελλοντικές γενναίες. Ο κύριος Αγγέλης δεν βρίσκεται εδώ, γι' αυτό θα δώσω το λόγο απευθείας στην κυρία Μάνερ. Έχετε το λόγο, κυρία Μάνερ. Θα... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το πολύ σημαντικό έγγραφο που εκπώνησε. Η Ευρώπη αλλά και ολόκληρο ο πλανήτη χρειάζονται πρώτε ύλε. Εμεί από πλευρά μα χρειαζόμαστε και αυτή τη στρατηγική. Έχει επανειλημμένω λεχθεί αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ όλο ιδιαίτερω ε, στι ε, πρώτε ύλε που θα έχουν όλο και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για τι επόμενε γενιέ. Σα υπενθυμίζω ότι ήδη στην έκθεση αυτή έχει γίνει ιδιαίτερο αλόγος για τις σκανδιναβικές χώρες και το τι μπορούν να κάνουν. Αν δει όλη την περιοχή της Αρκτικής που βρήθη πόρων, πολύ σημαντικών για το μέλλον, η Κομισιόν από δική της πλευράς ίσως θα έπρεπε να διευκρινίσει κάπως τα πράγματα. Ιδίως όταν κάνει λόγο για τους πόρους οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρώπη και όταν μιλά για την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Και βέβαια όταν μιλά και για τις σχέσεις με τρίτες χώρες. Ελπίζω χάρη στη στρατηγική αυτή να μπορέσουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας, ιδίως ό,τι αφορά τα πολύτιμα μέταλλα. Χαίρομαι που επετέχθη συμφωνία στο θέμα της φορολόγησης αυτών των σπάνιων πολύτιμων μετάλλων. Ελπίζω να μπορέσουμε τις πρώτες ύλες να τις εξοπίσουμε με καλύτερο τρόπο. Και θέλω να επιμείνω στο πόσο σημαντικό είναι το έγγραφο αυτό για τις επόμενες γενιές. Βέβαια, με απογοητεύει λίγο το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί απαρκώς υπόψη στο θέμα των δασών. Ενώ για την πράσινη οικονομία η δασοκομεία έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάνερ. Επόμενη ομιλήτρια κυρία Ντελάγκε. Eh, er Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε μια στοχευμένη πολιτική για τις πρώτες ύλες, ε, συγκεκριμένα για το το φόσφορο που είναι απαραίτητο για την ε, γεωργία και τα ε, παγκόσμια αποθέματα έχουν, είχαν εξαντληθεί πριν από πέντε χρόνια ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ο, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 9 δίσε που θα θέλουν, ε, περιμένουν να φάνε από αυτές τις καλλιέργειες. Πρέπει να αφήσουμε πια τα ευχολόγια και να περάσουμε στη δράση εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να βρούμε ε, ουσίες αντικατάστασης, να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μειώσουμε την επιβάρυνση για το περιβάλλον και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα, τις ουσίες που μπορούν να αντικαταστήσουν ε, πρώτες ύλες που έχουν κλείψει. Θα συμφωνήσω με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια που ε, προορίζονται για την ε, πρασινοποίηση σε εισαγωγικά της ε, οικονομίας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά τεχνικό το ζήτημα, αλλά δεν χρειάζεται να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι θα πρέπει χωρίς να το πολυσκεφτούμε να περάσουμε στη δράση και κυρίως να είμαστε ρεαλιστές όταν ε, χαράξουμε την μελλοντική πολιτική μας. Ελπίζω να αναλάβει συγκεκριμένη δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, πότε μπορούμε να αναμένουμε πρόταση από πλευρά σας, Πρόεδρος, η κυρία Τικάου. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή που ε, ενσωμάτωσε στην έκθεσή του τις τροπολογίες που καταθέσαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τις εισαγωγές πρώτων υλών και η ζήτηση για τις ε, πρώτες ύλες θα είναι συνάρτηση των αποτελεσμάτων των λαϊκών εξηγέσεων στις αραβικές χώρες και άλλων διεθνών εξελίξεων. Ε, η ζήτηση και η προσφορά είναι πράγματα που αποφασίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως δεν επικρατεί διαφάνεια σε σχέση με τις ε, ποσότητες ε, που εξορίζονται και τις ποσότητες των πρώτων που χρησιμοποιούνται για κάποια προϊόντα όπως τα κινητά τηλέφωνα. Ε, όπως για τους ε, με, ε, μεταλλάκτες, για τις οπτικές ίνες, για τους υπεραγωγούς, διάφορες διάφορα μεταλλεύματα που είναι απαραίτητα ώστε να είναι αποτελεσματική από οικολογικής πλευράς η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ρίνω τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα να ε, ε, εκπονήσουν ένα νέο πρόγραμμα καινοτομία με στόχο να αντικαταστήσουμε τις πρώτες ύλες ε, που δεν έχουμε σε επαρκή ποσότητα. Επίσης, ανακύκλωση. Πολύ σημαντικό, διότι ε, η ανάκτηση πρώτων υλών από τα απόβλητα, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση είναι μέτρα φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά μόνο αν γίνονται με σωστό τρόπο, αλλιώς είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Στην Αυστραλία, την Ασία, την Ινδία, το Μερκοσούρ υπάρχουν αντίστοιχοι προβληματισμοί. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Ινδία και η Βραζιλία στην 5η Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Βραζιλίας ε, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Αυτό θα είναι ένα ε, ζήτημα κέρια σημασίας συνδέεται με την ίδια την οικονομική ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να ελοποιήσει αυτά που υπόσχεται στην αρχική της πρόταση. Ευχαριστώ. Περνούμε στον επόμενο μιλητή, τον κύριο Φλόρενς. Ε, αγαπητέ Ράινχαρτ Μπιουτικόφερ, σε ευχαριστώ θερμά από αυτή τη θέση για την καλή και ισορροπημένη σου έκθεση. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την έκθεση και πιστεύω ότι αυτή η έκθεση θα συμβάλλει ούτε ώστε το πρόβλημα συνείδησης που έχουμε στην Ευρώπη, συνειδητοποίησης, ε, τεθεί. Ε, ξέρουμε πόσο περιμέναμε αυτή την έκθεση και το φτάξιμο δεν ε, βρίσκεται στον Ταγιάννη αλλά σε όλους τους, και σε όλους τους συνεργάτες του. έχουμε την πληροφορία από το τελευταίο Συμβούλιο Περιβάλλοντος ότι ο Πίτροπος παρουσίασε τη στρατηγική για τις πρώτες ύλες και υπήρξε ομόφωνη στρατηγική, λεκτικά επεφρασμένη για αυτή την έκθεση. Και μετά ήρθαμε στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης Electric Rays ε, ε, ε, οδηγία και χάθηκε κάθε ομοφωνία όταν το ζητούμενο ήταν να διατυπωθούν συγκεκριμένα μέτρα. ήταν μια πραγματική κοιλάδα των δακρύων. Το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με την Κομισιόν. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τη στάση του κυρίου Ποτότσνικ πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα φέρει κάποια κίνηση σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί ε, αν το πρόβλημα του κλίματος είναι μόνο κατ' τόσο σοβαρό ε, όπως ακούμε, τότε χρειαζόμαστε εξαιρετικά καινοτόμε υπήρους όπως είναι η Ευρώπη που θα αναπτύξουν ε, προηγμένες τεχνολογίες σε σχέση με τις πρώτες ύλες. Πιστεύω ότι οι τρεις πυλώνες που πρότεινε η Επιτροπή ε, και ίσως θα πρέπει να ακολουθεί η σειρά αυτή και εδώ διαφορούμε από τους πράσινους συναδέλφους νομίζω θα πρέπει να ρυθούν από κοινού και όποιο θέλει να ερμηνεύσει με κακό βουλοτρόπο την διπλωματία των πρώτων υλών μπορεί να το πράξει. Εγώ θεωρώ ότι το ζητούμενο εδώ είναι να έχουμε μια σωστή ε, ε, δίκαιη στάση έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών ούτως ώστε να βρούμε ένα τρόπο αντιμετώπισης ε, ώστε οι περιοχές αυτές να υποφελούνται από αυτές τις αριστηριότητες και να μπορούν να οικοδομήσουν σχολεία για παράδειγμα. Ε, το τρίτο σημείο έχει εξή. Υπάρχουν σημαντικέ ευκαιρίε για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, γιατί πρόκειται για την υποκατάσταση πρώτων υλών που θεωρούμε σήμερα ότι είναι φυσικέ, όπω είναι για παράδειγμα ο χαλκό. Ε, και μελλοντικά οι χάλκινοι αγωγοί θα ανήκουν στο παρελθόν και θα έχουμε νέα υλικά για τους αγωγούς αυτούς. Εδώ βρίσκεται ένα σημαντικό δυναμικό για την ε, βιομηχανία. Η ΕΦΕΦΑ είναι καλή. Η οδηγία αυτή είναι καλή, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ε, εξ ολοκλήρου σαν προστασία του περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να γίνει όπλο κατά της ε, πολιτικής των πρώτων υλών. Ο τρίτος ε, πυλώνας είναι σε συνάρτηση με το τι θεωρούμε εμείς στην ευρωπαϊκή πολιτική ως αποτελεσματική πολιτική ανακύκλωση. Εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλόρεντς. Ο, κύρι, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σταμπάζδη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίθεται το θέμα των πρώτων υλών σαν θέμα μείζωνο σημασία. και ήταν κατόπιν δική μου πρωτοβουλία συμπεριλήφθηκε εδώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μπιτικόφερ που ασχολήθηκε με τη μεγαλύτερη πρόκληση του 21ου αιώνα. Η έκθεση αυτή πραγματικά ασχολείται με το θέμα αυτό εις βάθος και με την ουσία του θέματος. Δηλαδή ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανακύκλωση των πρώτων υλών. Στο Ισραήλ Ε, είναι 70% στην Ευρώπη είναι μόνο 25% αυτό το ποσοστό. Δεν θα πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες όσον αφορά την ε, ανακύκλωση των ε, αποβλήτων. Όταν συνέβη στην Ουγγαρία το ατύχημα με την κόκκινη λάσπη, οι θύνοντες συζήτησαν σχετικά και τέλος οι βιομήχανοι κατέληξαν στο αποτέλεσμα ότι η ανακύκλωση θα ήταν ιδιαίτερος δαπανηρή στην περίπτωση αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Στόλογεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους άλλους συναδέλφους μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οποίοι έχουν ε, συμβάλει στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, έναν όλο και αυξανόμενο ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τι πρώτε ύλες. Ανταγωνισμό που θα γίνει όλο και πιο επιθετικό στο μέλλον λόγω του ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την πληθυσμιακή αύξηση στις αναψώμενες χώρες αλλά και να κατανοήσουμε ότι υπάρχει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας επίσης στις αναπτυσσόμενες αυτές χώρες. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης σε πρώτες ύλες. Επίσης, ε, ο γεωγραφικός εντοπισμός ε, σε συγκεκριμένες περιοχές και χώρες των πρώτων υλών περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες τείνουν να χρησιμοποιήσουν ε, πολιτικά για πολιτικούς σκοπούς τις πρώτες που διαθέτουν. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι κυβερνήσεις αρκετών χωρών έχουν βιομηχανικές πολιτικές οι οποίες στηρίζουν τις ντόπιε εταιρείε στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού. Και δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε ότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται και δημόσια κονδύλια για την δημιουργία πλεονεκτήματος για τις ντόπιε εταιρείε. Και πρέπει να αναλάβουμε δράση με ικανοποιεί η στρατηγική και η κατεύθυνση που έχει πάρει. Πρέπει να αποσυνδέσουμε την ενεργειακή απόδοση από τις πρώτες ύλε. Τώρα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τις ευρωπαϊκές εταιρείες και αυτό πρέπει να το κάνουμε με πολιτικές οι οποίες ευνοούν τη δημιουργία στρατηγικών συνασπισμών και την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε χώρες που είναι πλούσιες ε, σε ε, πρώτες ύλες. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ρόιλ, ο επόμενος ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, έγινε πολύ λόγος για τη σημασία των πρώτων υλών, για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πολλοί επεσήμεναν το πόσο μεγάλη είναι εξάρτηση των ε, επιχειρήσεων από τις ορυκτές ε, πρώτες ύλες. Ε, και το τελευταίο παράδειγμα ήταν η επισήμανση σε μια μικρή εταιρεία για λαμπτήρες όπου οι λάμπες αυτές είναι ιδιαίτερως δαπανηρές ε, ε, λόγω ακριβώς των σπάνιων γεών. Και είμαι ευγνώμων προς τον κύριο Μπιουτικόφερ, ο οποίος ε, κατάφερε να βρει μια ισορροπημένη απάντηση. Για παράδειγμα, ως προς το ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα, σημαντικό δεν είναι ο καθένας πάει το κεφάλι του και να παρουσιάζει τη δική του άποψη σαν ορθή, αλλά να υπάρξει μια συνεργασία. Και νομίζω ότι όσο αφορά την πρόταση της Επιτροπής για, τις τρεις, για τους τρεις πυλώνες, ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το πώς μπορούμε να έχουμε πρώτες ύλες στην Ευρώπη. Ο συνάδελφος κ. Ε, Φλόρεντς επεσήμανε τις αντιφάσεις με τις άλλες νομοθεσίες και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα όρια τι επιθυμούμε εμείς, πώς μπορούμε να ε, έχουμε πρώτες ύλες ναι, από θέματα πρώτων υλών στις πρώτες στην Ευρώπη. Ε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε με την ανακύκλωση. Αλλά θα πρέπει να δούμε και το θέμα της οικονομικότητας. Η, τώρα, η διπλωματία των πρώτων υλών. Αναφέρθηκε σε αυτήν ένα συνάδελφος σαν ένα εργαλείο που θέτει τους άλλους υποπίεση. Αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι μια παρανόηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικές οι διεθνείς ε, συζητήσεις ούτως ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε το δικό μας δυναμικό εδώ στην Ευρώπη και ε, βεβαίως θα πρέπει να έχουμε ένα σωστό τρόπο στη μεταχείριση των άλλων χωρών. Η Κομισιόν ε, το να λέμε ότι η Κομισιόν μας υπαγορεύει τη χρήση των πρώτων υλών, θεωρώ ότι αυτό είναι εσφαλμένο. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να εξασφαλίσουν ότι παραμένει η διατύπωση ως έχει της έκθεσης αυτής για να μπορέσουμε να την ε, υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει και προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες ε, σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες. Η πρόκληση βασικά, οι προκλήσεις πρέπει να γίνουν ευκαιρίες για να βελτιωθεί η βιομηχανική ισχύ τη Ευρώπη, Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική καινοτομία για την αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών στην Ευρώπη. Γιατί κάτι τέτοιο θα συμβάλλει στην υψηλότερη ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα αλλά και στην ε, ασφάλεια των εφοδιασμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνάψει εταιρικέ σχέσει με τρίτε χώρε αλλά και να σταθεροποιήσει ε, τι ε, διαπραγματεύσει και ρυθμίσει ό,τι αφορά τι πρώτε ύλε. Πρέπει να υπάρξει μια διεθνή πλατφόρμα για να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτε ύλε από τρίτε χώρες. Θα πρέπει να τονίσουμε την εξάρτηση τη ευρωπαϊκή βιομηχανία από τι πρώτε ύλε και θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε τι σημερινέ και μελλοντικέ τιμέ των πρώτων υλών. Αν γίνει με τέτοια μελέτη, θα μπορέσουν και τα κέντρα ερευνών να κάνουν ε, μακροχρόνιε επενδύσει. Περάσουμε τώρα στην ε, διαδικασία προσέλκυση τη προσοχή του Προέδρου Catch the Κυρία Μαγκίνε, βλέπω ότι θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Σιγητά, θέλω να σα ευχαριστήσω για την εκθέσή σας, η οποία με ευρυτέρα ταινία μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Μιλάμε για συγκεκριμένες πρώτες και θέλω να συμφωνήσω με τα σχόλια της κυρίας Ντελάγκε για το φωσφόρο και για το ότι μειώνονται τα αποθέματά του. Και θα πρέπει να ξαναδούμε το πώς θα μπορούμε να παράγουμε τρόφιμο, όχι μόνο εντός ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντα υπόψη ακριβώ και αυτό το ε, συστατικό, το φωσφόρο που είναι τόσο σημαντικό για τα τρόφιμα. Η έκθεση έχει λάβει υπόψη και κάποια σχόλια τη Επιτροπή Γεωργία. Ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά την προσέγγιση των τριών πυλώνων, δεν μιλάει για γεωργία και τρόφιμα, αλλά για κάποια άλλα κεκτημένα και κάποιου άλλου κλάδου. Αυτό είναι σφάλμα κατά την άποψή μου, γιατί ένα από του πιο κρίσιμου τομεί, κατά την άποψή μου, για τον κόσμο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η ασφάλεια των τροφίμων και χρειαζόμαστε πρώτε ύλε για την παραγωγή τροφίμων. Πολλά από αυτά τα οποία έρχονται στην ε, τροφική αλυσίδα είναι σπάνια ε, και θα πρέπει να ε, φροντίσουμε να συνεχίσει να υφίσταται υφίσταται γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μακγκίνες. Επόμενο μιλήτρια τώρα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την, ε, πολύ, για την πολύ καλή σας εργασία. Εδώ έχουμε πάρα πολλούς ε, κινδύνους, ε, οι τιμές που δεν είναι προβλέψιμες καθώς και ανταγωνιστικότητα. Και εδώ θα πρέπει να δούμε την, τη χρήση της, των ευρωπαϊκών φυσικών πόρων. Θα πρέπει να έχουμε μια αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών. Η οικολογική αποτελεσματικότητα θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, ούτω ώστε οι πόροι να μπορούν μέσω τη ανακύκλωση να χρησιμοποιούνται, πολλέ πολλές φορές. Η ανακύκλωση είναι ιδιαίτερο σημαντική εδώ. Θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω την πρόκληση της Επιτροπής να χαράξει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα μέχρι το 2050 για τις πρώτες ύλες. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Μέλτσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι για παράδειγμα σε ένα κινητό γνωστά μέταλλα όπως ε, χαλκός περιέχονται αλλά και λιγότερο γνωστά μέταλλα ε, τα οποία θα είναι αναγκαία για τις μελλοντικέ τεχνολογίες. Ε, και λόγω της εξαγγελίας της Κίνας ότι 97% των, το βάρη των 7% των μετάλλων θα πρέπει να κινηθούμε ε, σύντομα και θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια βιώσιμη στρατηγική στην Ευρώπη και θα πρέπει να σκεφτούμε ακριβώς ε, ποιες είναι οι δικές μας ανάγκες που θα πρέπει να, ε, να καλύψουμε άμεσα. δεν θα πρέπει η ανακύκλωση ε, λόγω των ε, σωρών αποβλήτων ε, είναι ιδιαίτερως ε, σημαντική. Αλλά δεν μπορεί να έχει, αποτελεί μια ριζοσπαστική λύση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μέλ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευτυχώς που εστιάζουμε σε αυτό το θέμα σήμερα, διότι ε, χωρίς μια λογική, εξορθολογισμένη στρατηγική για τις πρώτες ύλες, αποκλείεται να σημειώσουμε πρόοδο. Ακόμη κι αν είστε ο καλύτερος ε, διαχειριστής στον κόσμο, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα αν δεν έχετε τις πρώτες ύλες. Και το ίδιο συμβαίνει και στη βιομηχανία. Θα πρέπει λοιπόν ε, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και σωστή έκθεση του κυρίου Μπίτι Κόφερ γιατί είναι κέρυες ε, σημασίας να έχουμε έναν πάγιο εφοδιασμό σε πρώτες ύλε για να είμαστε ανταγωνιστικοί και πρώτα πρέπει να στραφούμε στις πρώτες ύλε που έχουμε εντός των συνόρων μας ε, και να μην παρεμποδίζουμε την ανάπτυξή τους με υπερβολικούς ε, περιορισμούς όπως είδαμε στο παρελθόν. Θέλουμε να είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς, αλλά δεν μπορούμε παρά να ανακυκλώσουμε. Η ανακύκλωση από πολλές πλευρές βρίσκεται σε παιδική ηλικία και ε, τα υλικά που ανακυκλώνται μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές. Οπότε ε, χρειαζόμαστε με αυτό το σύστημα λιγότερες βασικές προτεσίλες. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ε, οι σπάνιες γιές έχουν κέρια σημασία και το 97% των σπάνιων γιών, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ε, χρησιμοποιούνται σε τόσες πολλές διαφορετικές ε, συσκευές ε, που πρέπει να μας απασχολεί το θέμα. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, να γίνουμε ανταγωνιστικοί και χάρη σε αυτή την πολιτική θα το καταφέρουμε συγχαρητήρια προ τον εισηγητή. Σα ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Η κυρία Ντανσίλα έχει ζητήσει επίση το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. όλοι ξέρουμε πώς ε, έχει με μεγάλες ευκαιρίες αλλά και πολύ μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των πρώτων υλών. Ε, αυτός ο τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το, τη βιομηχανία και το διεθνές εμπόριο αλλά ταυτόχρονα αφορά και σε οριζόντιες ε, πολιτικές για την εσωτερική αγορά αλλά και για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία αποτελεσματική εποπτεία της εφαρμογής των πολιτικών είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία αυτών των πολιτικών. Επίσης χρειάζεται στενότερο, ε, αποτελεσματικότερο συντονισμό ανάμεσα στη δράση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτός ο εποπτικός ε, μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει και στο Κοινοβούλιο να βλέπει ακριβώς ε, τι συμβαίνει, να προβλέπεται μια ετήσια έκθεση, μια ετήσια αναφορά. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστούμε κυρία Ο Κύριος Ρώση, παρακαλώ. Ταγιάννη, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η μείωση της κρίσης ε, πρώτων υλών έχει πολλά πλονεκτήματα και από πλευράς περιβαλλοντικής, περισσότερη ανάκτηση, λιγότερα απόβλητα και μικρότερη επιβλαβής ε, επέμβαση στο περιβάλλον. Πρέπει βέβαια να γίνουν τα απαραίτητα σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό. Γι' αυτό και οι διάφορες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται Διεθνώ και πρέπει να αναλάβουμε όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο τι ε, απαιτούμενε δεσμεύσει. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι θα πρέπει την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να την λάβετε υπόψη σα ε, την δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Αγορά ενέργεια που προωθεί και ο πρόεδρο Μπούζικ. Θέλουμε να έχουμε εφοδιασμό, ασφάλεια και για τι τιμέ. και θα εξοικονομήσουμε και σημαντικού πόρου. Ε, σημαντικό για την οικονομία, για τη βιομηχανία και τον πολιτισμό μα εν γέννη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπασέσκου. Μικρόφωνο παρακαλούμε γιατί σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αποτελεσματική στρατηγική για τις πρώτες ύλε εάν θέλει να παραμείνει από ποιομανική άποψη ανταγωνιστική. Μεταξύ των ουσιοδών παραμέτρων για τον ανταγωνισμό μπορούμε να συμπεριλάβουμε τη διπλωματία των πρώτων υλών που να είναι περιεκτική και αποτελεσματική. Και αυτό είναι τέλος σημαντικό γιατί η προμήθεια των πρώτων υλών επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία των διπλωματικών εργαλείων και διατυπώνει συγκεκριμένες υποδείξεις για τη συνεργασία με τους εξωτερικούς εταίρους. Για παράδειγμα, την υποστήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες συμπεριλαμβάνοντας ε, την ε, μεταφορά γνώσεων. Επίσης θα ήθελα να τονίσω την ε, σημασία του συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πολιτική των χωρών μελών. Και ελπίζω ότι η EEAS θα μεταποβεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Κυρία Μέρκης είναι τελευταία ομιλήτρια στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ. Θα ήθελα να πω τα εξής. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στην έκθεση της Επιτροπής και στη δική μας ε, έκθεση. Πρέπει επίσης ε, να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Ε, η αποθήκευση, δεν ξέρω, κάποιος την ανέφερε, αλλά δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο μέτρο. Επίσης, ε, πολύ λόγος έγινε για το φωσφόρο, για τα πρώτες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Σημαντικά είναι και αυτά τα θέματα, αλλά αυτό που με απασχολεί εμένα είναι πώς θα φροντίσετε να υπάρχει καινοτομία, περισσότερη καινοτομία στον τομέα αυτό. Έχουμε στόχους αποδοτικότητας ε, που τελικά δεν είχαμε, μάλλον αλλά βγήκαν την έκθεση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τις ε, επαναφέρουμε αυτές τις και για την κατάρριξη των αρκών ξηράς, για την καινοτομία και σε ό,τι αφορά τα απόβλητα νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ε, έχουμε μεγαλύτερη ανακύκλωση των αποβλήτων. Σε ό,τι αφορά τώρα το συντονισμό, πώς θα υπάρξει συντονισμός, ποιος θα οργανώσει, ποιος θα το κάνει εσείς ή ο κύριος Ποτότσνικ. Ευχαριστώ κύριο Σταγιάννη, ο Επίτροπος. Ακούσατε κύριε Επίτροπε όλα τα επιχειρήματα, όλα τα ερωτήματα. Είναι η ώρα να απαντήσετε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επαναλάβω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατά τη γνώμη μου συνάδει πλήρως με την έκθεση του κυρίου Μπιτικόφερ. Εμείς ε, ποντάρουμε σε μία στρατηγική ως προς τις ε, πρώτες ύλες, μια στρατηγική που θα ε, είναι ισοβαρής, ισορροπημένη και θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες, ε, την εσωτερική στρατηγική που θα εφαρμόζεται δηλαδή στην επικράτεια της Ένωσης, την εξωτερική στρατηγική της Ένωσης και ε, τη δράση μας υπέρ της καινοτομίας. Και θα αρχίσω από αυτό το τελευταίο στοιχείο. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια εξισορροπημένη στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα από τα αρχικά της ε, ε, έγγραφα για αυτό το θέμα τόνισε τη σημασία των εταιρικών σχέσεων, στρατηγικής σημασίας. Ε, λάβαμε την ε, σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και έτσι θα προχωρήσουμε με την προσήλωση και τη συνεργασία ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια εταιρική σχέση για την ανακύκλωση. Δεν είναι σε καμία περίπτωση υποδέστερη αυτή η εταιρική σχέση. Δηλαδή, προτού εκπονηθεί το έγγραφο για τις πρώτες ύλες, μιλήσαμε για την εταιρική σχέση, για την ανακύκλωση και ε, σε πρώτα ε, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει αυτήν την εταιρική σχέση και μετά ασχολήθηκε με τι πρώτες ύλε. Ε, και δεν καταλαβαίνω γιατί απουσιάζουν οι βουλευτές που έθεσαν τα σχετικά ερωτήματα. τέλο πάντων εμείς ταχθήκαμε υπέρ τη επαναχρησιμοποίηση και τη ανακύκλωση και αυτή μα η απόφαση προηγήθηκε της δημοσίευσης τη έκθεση για τι πρώτε ύλε ω προ την στρατηγική που θα εφαρμοστεί στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε, ίσως ε, δεν ε, κατάλαβα ε, ακριβώς το ερώτημά σας ή δεν καταλάβατε εσείς την αρχική μου παρουσίαση. Εγώ μίλησα για τη Γρυλανδία διότι η Γρυλανδία είναι μία από τις χώρες που θα επισκεφτούμε για να εργαστούμε, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα των πρώτων υλών. Συμμετείχαμε τη Σουηδική κυβέρνηση σε ένα θέμα το οποίο οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο προέδρευε και ο Υπουργό Εξωτερικών τη Σουηδία και αναφερόταν σε πρωτοβουλίε για πρώτε ύλε στη θάλασσα του Μπάρεντ. Μίλησα και με τον Υπουργό Εξωτερικών και έχουμε επιβεβαιώσει μια επίσκεψη για να πάμε να δούμε επιτόπου τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τι πρώτε ύλε. Σα το λέω αυτό διότι. Ε, μίλησα Ιταλικά και μπορεί να υπήρχαν κάποιες ανακρίβειες. Ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω κύριε Πουσκόη, δεν την ξέχασα τη Σουηδία. Η Γρυλανδία άλλωστε ήταν ε, τμήμα της Δανίας μέχρι πρόσφατα. Και τώρα υπάρχει μια ε, ένωση με τη Δανία, επομένως δεν απέχει και πάρα πολύ από την σχέση με την Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα τη διεθνή πολιτική, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση και λυπάμαι που δεν είναι στην αίθουσα αυτή τη στιγμή η κυρία Ματίας και Φιγκερέιδο, δεν έχω καμία πρόταση, πρόθεση συγγνώμη, να ακολουθήσω νεοαπικιακές πολιτικές στην Αφρική. Προέρχομαι από μια χώρα η οποία ήταν η πρώτη χώρα που ζήτησε συγγνώμη από την Αφρική για τα σφάλματα τα οποία διαπράχθησαν στη διάρκεια της και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει νεοαπικιακή πολιτική στη συγκεκριμένη Ήπειρο. Ιδιαίτερα για το θέμα των πρώτων υλών, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή, έντονη συμμετοχή των Αφρικανικών χωρών και όλα αυτά συζητήθηκαν με την Αφρικανική Ένωση σε στενή επαφή με πολλές χώρες της ε, Αφρικανικής Ένωσης διότι η Αφρική δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί θύμα της νέας αποικιοκρατίας. και σε καμία περίπτωση δεν είναι η Ευρώπη αυτή η οποία έχει αποικιοκρατικές τάσεις αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα ένα θέμα το οποίο υπευλήθη στη διάρκεια της παρουσίασης της γνωμοδότησης το, από τον κύριο Σνίμπερ, Νάγκε και υπογραμμίστηκε και από την κυρία Εκ. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για τη διαφάνεια των εξορρυκτικών βιομηχανιών και αποτελεί αναδυόμενη δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο για τις ευθύνες ε, του κλάδου. Εντατικοποίησαμε τις προσπάθειές μας για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και στο σχετικό ταμείο έδωσαν συγχρηματοδοτήσεις ε, για συνεδριάσεις επιρρογνωμόνων, για συμμετοχή μεγαλύτερη από πλευρά Συμβουλίου. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ελλείψεις ακόμα, οι οποίες απορρέουν από το γεγονός ότι ε, πέραν που 50 χώρες ε, συμμετέχουν, αλλά μόνο 9 μέχρι τούδε τηρούν τους κανόνες ε, της πρωτοβουλίας της εξορυκτικής βιομηχανίας. Όσον αφορά τώρα την επίσημη πρόταση που θα πρέπει να παρουσιαστεί όσον αφορά την υποχρέωση των χωρών, μετά από συζήτηση με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρχει υποχρέωση λογοδοσία σε χρηματοοικονομικό επίπεδο για τις επιχειρήσεις ε, ε, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε στα πλαίσια ε, του επόμενου έτους να παρουσιάσουμε μία νομοθετική πρόταση. Και θέλουμε να ενισχύσουμε τα θέματα της διαφάνειας και θα τα λάβουμε υπόψη με το, υπό το ίδιο πνεύμα του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μπουτικόφερ. Η συζήτηση και η διαβούλευση έγινε από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι το 2011 και αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση. Όσον αφορά τώρα το τελευταίο ζήτημα, αυτό το οποίο ετέθη όσον αφορά το θέμα της αποθήκευσης, θεωρούμε ότι το να διασφαλίσουμε την διαθεσιμότητα πρώτων υλών για τις επιχειρήσεις είναι ρόλος των ε, θεσμικών και πολιτικών αρχών και θα πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης και τις ιδανικές συνθήκες εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως είναι διατεθειμένη να συζητήσει σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα ενός προγράμματος αποθήκευσης πρώτων υλών, το κατά πόσον είναι υλοποιήσιμο και εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το υφιστάμενο σύστημα για την αποθήκευση πετρελαίου. Ε, ξεκίνησε και μία διερευνητική εξέταση η οποία είναι ακόμα εν εξελίξη. Δεν απάντησα σε όλα τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν στη διάρκεια της συζήτησης, αλλά εάν απαντούσα αναλυτικά σε όλους θα έπρεπε να μιλήσω άλλη μισή ώρα. Καλύτερα θα ήταν να ακούσουμε τον κύριο Μπουτικόφερ. Είμαι όμω στη διάθεση όλων των Ευρωβουλευτών για να συζητήσουμε ακόμα και διμερώ όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ε, κοινοτική στρατηγική σε θέματα πρώτων υλών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τον τελευταίο λόγο δίνω στον κύριο Μπιτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλες και όλους για τις παρεμβάσεις σας καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ταγιάννη για τις παρατηρήσεις ε, που συνέβαλε, καθώς επίσης και για την υποστήριξή του υπέρ ενός δικτύου αρμοδιοτήτων, καθώς και για τις άλλες προτάσεις που έκανε στην πράξη. Μιλήσαμε πολύ για την εξόριξη πρώτων υλών. Ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνουν. Ωστόσο, ιδίως σε οικολογικά ευαίσθητε περιοχές πρέπει να προχωρήσουμε και με ιδιαίτερα ευαίσθητο τρόπο. Είναι σημαντικό, αυτό το λέει άλλωστε και η έκθεση, να μην προκαλέσουμε καμία εσφαλμένη αντίθεση ανάμεσα στη βιομηχανική πολιτική και στην προστασία του περιβάλλοντο. Και γι' αυτό με ικανοποίησε άκουσα ότι οι γενικέ σα διευθύνσει περιβάλλοντος και επιχειρήσεων μπόρεσαν τελικά να συμφωνήσουν. Τα ορυχεία μας είναι και τα παλαιά ας πούμε εργαλεία τα οποία έχουμε ακόμα στα συρτάρια μας. Επίσης η ανακύκλωση πρέπει να γίνει ένα οικονομικό μέσο, ένα οικονομικό εργαλείο. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινιάστηκε η πιο σύγχρονη στον κόσμο εγκατάσταση ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου. Το απόρριμα πρέπει πλέον να αντιληφθούμε ότι είναι ένα σύγχρονος τρόπος Ανάκτηση πρώτων υλών. Πρέπει να συνεχίσουμε να τα συζητούμε αυτά τα πράγματα. Ακούω από ορισμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφορετικέ φωνέ. Γνωρίζω ότι ο Επίτροπος κ. Ντεγκούχτ, για παράδειγμα, τηρεί επικριτική στάση. Δεν ξέρω πώ θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, για παράδειγμα, για τι σπάνιε γέε, όταν βλέπουμε την Κίνα να περιορίζει ακόμη την παραγωγή. Για την κυρία Γκέρλινγκ, η οποία είναι απούσα τώρα, θέλω να πω ότι πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά και βεβαίως με μελέτες επιπτώσεων. Εν τέλει, για τα εξωτερικά, για μένα η πολιτική πρώτων υλών δεν είναι νέο απεικιοκρατία. Η ΔΕΜΗ, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο δεν θα αναγνώριζαν την αρχή της κυριαρχίας επί των πρώτων υλών. Και αν με επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε να πω μια φράση